της ημερήσιας διάταξης. Έχουμε τρία σχέδια ψηφίσματος για την Ικαράγουα και θα δώσω το λόγο στους ε, εισηγητές. Συντάκτες των ψηφισμάτων, πρώτος ο κύριος Μπογκούσο Αφασόνικ. Πολιτικά. Ευχαριστώ. Η πολιτική του Δανιέλ Ορτέγκη, του ισχύοντος του ενεργεία Προέδρου της Νικαράγουας, είναι η νοοτροπία της παλιάς κομμουνιστικής ε, ιδεολογίας από τη στιγμή που, κρατάμε, που λαμβάνουμε την εξουσία δεν την αφήνουμε από τα χέρια μας. Και μετά την, τους ε, η Νικαράγουα χρειάστηκε να αποδεχθεί τους κανόνες του δημοκρατικού παιχνιδιού και μάλιστα το 2006 ε, ο Ορτέγα επανήλθε στην εξουσία, οι σαντινίστες ανέλαβαν και πάλι τα ενία και άρχισαν ε, με ψευδονομικίστικους ε, στόχους να προσπαθούν να εξαλείψουν την αντιπολίτευση. Και μάλιστα κυριάξαν σε όλα τα επίπεδα της εξουσίας. Μάλιστα πριν από λίγα χρόνια εμείς ε, ε, επισημάναμε τον κίνδυνο ε, προσπάθειας ε, εξαφάνισης της αντιπολίτευσης, εκφοβισμού και δίωξης των δημοσιογράφων, ε, φήμωσης ε, του τύπου και μάλιστα πολλά διεθνείς οργανώσεις επισήμαναν αυτό το θέμα και η χειραγώγηση του Ορτέγκα οδήγησε σε αλλαγή του συντάγματος ε, προκειμένου να παραταθεί η θητεία του και νομίζω ότι το επόμενο βήμα του θα είναι να ανακηρυχθεί Σόβιος πρόεδρος. Μάλιστα πρότυπο ηγέτη για τον Ορτέγα είναι ο Φιτελ Κάστρο. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε αυτό το θέμα και στην καταστρατήγηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που γίνονται στην Ικαράγουα. Μήπως θα έπρεπε να αναστείλουμε τις συμφωνίες που έχουμε με τη χώρα αυτή μέχρι ότου να εφαρμοστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα γιατί, για να μην μείνουν κενό γράμμα όλες οι εκκλήσεις που κάνουμε για, την, για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο κύριος Μπιέλαν, ευχαριστώ. Την περασμένη, το περασμένο Σάββατο δεκάδες χιλιάδες ε, υπήκοοι πολίτες της Νικαράγουας ε, διαμαρτυρήθηκαν μετά από έκλεισε της αντιπολίτευσης κατά του Προέδρου Ορτέγα. Γιατί ο πρόεδρος αυτός επιχειρεί να ε, επαναφέρει τη δικτατορία στην Νικαράγουα. Και μάλιστα θυμάστε τον Οκτώβριο τι έγινε με την προσπάθεια παράτασης της προεδρικής του θητείας. Τέτοιου είδους απαγόρευση υπάρχει σε ευρωπαϊκές χώρες, αλλά ε, βέβαια ο Ορτέγα δεν έχει τα, την πλειοψηφία των δύο τρίτων στη Βουλή. Γι' αυτό χρειάστηκε για να καταργήσει αυτή την απαγόρευση παράταση τη θητεία ε, να προτείνει μεταρρύθμιση του συντάγματος. Νομίζω ότι είναι εξοργιστική η κατάσταση που επικρατεί στην Νικαράγουα που ισοδυναμεί με μια πραγματική δικτατορία. Γι' αυτό απευθύνομαι στην ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε στις επόμενες διαπραγματεύσεις ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες Κεντρικής Αμερικής να επισημάνει αυτό το πρόβλημα της Νικαράγουας και να ε, χρησιμοποιήσει κάθε μέσο προκειμένου να ανατρέψει τις προθέσεις του Πρόεδρου Τέγκα. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Βαμπάλεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι θα ευγνώμονες προς το Κοινοβούλιο την Αντιπροσωπεία και την Αποστολή στην ε, Μανάγουα. Για το Σύνταγμα, για τις εκλογές, για την προεκλογική εκστρατεία, τις ε, πολιτικές ελευθερίες, τα ανθρώπινα δικαιώματα, όλα αυτά εκεί τα, τα, τα, τα προωθήσαμε και μας απειλήσανε persona non grata θέλανε να μας ε, κηρύξουν κάτι σαν πραξικόπημα. Παρ' όλα αυτά όμως καταδικάζεται έτσι. Η χώρα αυτή σε μια κατάσταση καταπίεση του λαού της όπου θα πρέπει όμως οπωσδήποτε η Ευρωπαϊκή Ένωση να στείλει αντιπροσώπους, παρατηρητές στις εκλογές για να βοηθεί το έργο της δημοκρατικής αντιπολίτευσης και ελπίζουμε ότι το αποτέλεσμα θα είναι κάτι που να αντιστοιχεί σε δίκαιες, ελεύθερες εκλογές. Και τελικά να γνωριστεί ότι έγιναν τέτοιου είδου ε, δίκαιε εκλογέ και έτσι να μπει τέλο στην κρίση μα τη χώρα. Ευχαριστούμε κύριε Φανμπάνη πρόεδρο Και τώρα οι αγορητέ των πολιτικών ομάδων. Πρώτο ο κύριο Κέλαμ για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στη Λατινική Αμερική υπάρχει μια σχετική τάση ότι δηλαδή κάποιες λαϊκίστικες κυβερνήσεις ε, παραμένουν ε, στα πράγματα και, και παρατείνουν οι επικεφαλείς τους την, την, την παραμονή τους ε, στην εξουσία. Το ίδιο ακριβώ έκανε και ο Χίτλερ, ο Λένιν. Όμως ε, τελικά έχουμε μία από τα ίδια. Οπότε βλέπουμε ότι αυτοί οι πρόεδροι με τις ιδιαίτερα διαβριμένες αρμοδιότητες δεν έχουν κανένας είδους έννοια για, για τους πολίτες τους. Να, είδατε τι έγινε στην Κούβα, πώς τσακίστηκαν οι ζωές των ε, ανθρώπων εκεί των απλών επί δεκαετίες στη Δένη Καράγουα. Πάλι βλέπουμε κάτι το πάρα πολύ ανησυχητικό. Είδαμε ότι και εκεί έχουμε μία από τα ίδια. Οπότε αυτό που είναι δικό μας ε, καθήκον είναι να καταδικάσουμε αυτές όλες τις ε, ατασταλείς αντισυνταγματικότητες στην Ικαράγουα και θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει σε σχέση με τα χρήματα που δίνονται για αναπτυξιακή βοήθεια στην ΕΚΑΡΑΓΟ Και επίση είναι πάρα πολύ δυσάρεστο το ότι για αυτέ τι κατάφορε παραβιάσει του ΣΤΑΜ δεν έκανε τίποτα η Αμερική. very much, Mr. Kalam. Κύριε Κελάμ, σα ευχαριστούμε, λέει ο πρόεδρο. Κύριε Αντεκάζη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε πρόεδρε. μεγάλη μου χαρά βλέπω ο κύριο Μπάλε γύρισε. Μπήκε στο αεροπλάνο για να επιστρέψει. Τι θέλω να πω. Πιο σοβαρά ότι είπα, είπαμε στην πολιτική μας ομάδα δεν θέλω να παίξουμε αυτό το παιχνίδι και άπαξ και το ΑΛΚ αρνήθηκε εκείνο το κατεπήγον θέμα για την Ουγγάντα και τους ομοφιλόφιλους επίσης καταψήφισαν ένα άλλο κατεπήγον που αφορούσε κάποιες εκτελέσεις στο Ιράν τώρα ξαφνικά θέλουν να μπούμε εμείς στο παιχνίδι σε σχέση με το, τα εκεί στην Ιχαραβού. Εγώ όμως δεν θεωρώ ότι εδώ τα κατεπήγοντα τα οποία πραγματικά αποσκοπούν στο να βοηθήσουν κάποιους ανθρώπους, κάποιες υποθέσεις ε, θα πρέπει να εξυπηρετούν κάποια πολιτικάντικα συμφέροντα κάποιων βουλευτών. Άρα, εμείς θεωρούμε ότι αυτού του είδους η πρόταση, αυτό το ψήφισμα είναι μια ντροπή για το Κοινοβούλιο. Ευχαριστούμε κύριε Δεκάζε, λέει ο Πρόεδρος. Ρωμέβα ή Ροέντα. Και εγώ πρεσβεύω τα ίδια. Είναι θλιβερό και είναι ντροπή το ότι έχουμε εδώ μια κατεπίγωσα συνεδρίαση η οποία ε, χρησιμοποιείται για να χειραγωγήσει τις εξελίξεις. Να, τώρα ας πούμε λέμε για την Ικαράγουα και σε άλλες περιστάσεις είχε γίνει το ίδιο, για ακόμα χειρότερες, πιο σοβαρές καταστάσεις. Και κάποια πράγματα που είναι στη μέση διάταξη διαγράφησαν. Οπότε, αυτό είναι πάρα πολύ κακό. Δυτική Σαχάρα, γιατί να μην μιλάγαμε. Η Αμινά Χαϊντάρ επίσης αυτή με υφίσταται στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων. Άλλοι, άλλοι πολλοί που βρίσκονται σε κατεχόμενα στο Μαράκο ή σε στρατόπεδα αχμαλώτων. Πρέπει επομένω να αποκτήσουν μια ξεκάθαρη θέση. Να, τι θα έπρεπε να σήμερα και τώρα να συζητούμε. Και δεν ξέρω γιατί το ΕΛΚ τώρα θέλει να συζητήσουμε για κάτι το οποίο ούτε έχει ενδιαφέρον, ούτε αξίζει ενδιαφέρον για τέτοιε ρυθμίσει. Ευχαριστούμε κύριε Ρωμεύα η Ρέδα. Και τώρα, για την ε, Ευρωπαϊκή Νοτιαστρία έχει το λόγο κύριε Φιγκέρετα. Είναι θλιβερή αυτή η συζήτηση, είναι ψευδοεπίγον το θέμα το οποίο εδώ επικαλούνται, είναι ε, ντροπή για το Κοινοβούλιο. Γιατί ας πούμε θα ήταν επίγον να πούμε τι έγινε με αυτόν τον τυφώνα, τον ε, κυκλώνα τον Νοέμβριο στη χώρα εκείνη. Κατέστρεψε τις υποδομές, κατέστρεψε νοσοκομεία, ε, υδραγωγία κλπ. Και τώρα καθόμαστε και λέμε τι θα γίνει με τα χρήματα σε σχέση με αυτό το κατεπήγον αντί να καθόμαστε και να λέμε πώς θα, βοηθήσουμε το Σαλβαδόρ. Και αυτό ήταν επίγον. Επίσης, το στρατηγικό πραξικόπημα στην Ονδούρα και αυτό ήταν ε, κατεπήγον με τον πρόεδρο Σελάγια. Βεβαίω και είναι κατεπήγον κάτι να γίνει για τα ανθρώπινα δικαιώματα για το, το, το λαό τη Δυτική Σαχάρα. Δυστυχώ όμω τίποτα από αυτά δεν γίνανε. Γιατί, γιατί ήταν κατά το Λαϊκό Κόμμα. Και όπως είπα και άλλοι συνάδελφοι, δεν πρόκειται να γίνουμε συνένοχοι αυτού του ψευτοκατεπήγοντος που είναι μια ντροπή για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο κύριο Κλούτε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να συμφωνήσω Καταρχήν με τους προλύσαντες. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι ο πρόεδρος της Κολομβίας προσπάθησε επίσης να παρατείνει την διάρκεια της θητείας κατά των ε, ισιών των νόμων της χώρας του. Θα πρέπει και αυτό να το συμπεριλάβουμε. Από την άλλη μέρα θα ήθελα να σας πω ότι το Ίδρυμα Friedrich Ναουμαν, που είναι πλησίον της FTP στη Γερμανία είχε συμμετάσχει στην εξέργηση στην Χοντούρα. Υπήρχε τουλάχιστον μια συζήτηση σχετική στην Γερμανία, υπήρχε μια ανοιχτή επιστολή σχετική. Ο κ. Βαλεν δεν μπορούμε να ξεχνάμε ότι είναι πρόεδρος της ε, Φιλελεύθερης Διεθνούς και στην ιστοσελίδα του αναφέρεται κάτι σχετικά με το πραξικό ε, Αυτό πρέπει να το... Να μην ξεχνάμε ότι είναι δικαίωμα της χώρας αυτής να απελάσει έναν άνθρωπο που αναφέρεται σε πραξικό μα σε μια χώρα. Η χώρα αυτή δεν χρειάζεται να τον υποδέχεται και θα πρέπει Νομίζω να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν ορισμένε κυβερνήσει στην ε, Λατινική Αμερική που προσπαθούν να ακολουθούν μια κοινωνική ε, πολιτική και έχω να σα πω ότι εμεί ε, δεν θα ακολουθήσουμε αυτή τη γραμμή, να του κατηγορούμε. Ευχαριστώ, λέει πρόεδρο. Τώρα έχουμε την διαδικασία Κατσουδιάη. Δύο λεπτά. Επειδή έχουμε πολλού όμω, εγώ θα δώσω το λόγο σε έναν ομιλητή από κάθε πολιτική ομάδα. Και θα αρχίσουμε με τον κύριο Κασουλίδη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πραγματικά δεν κατανοώ την αντίδραση των αξιότιμων συναδέλφων που κάθονται δεξιά, στη δεξιά πτέρυγα του Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά την επιλογή των σημερινών κατεπηγόντων. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν θεωρούν κατεπήγον να συζητήσουμε ε, το θέμα της μεταχείρισης ενός Ευρωβουλευτή που επισκέφθηκε τη χώρα αυτή ασκώντας ε, τα δικαιώματά του Προέδρου της Liberal International. Γιατί λοιπόν ε, να μην δικαιούμαστε το λόγο για να θίξουμε αυτό το θέμα και επίση να μιλήσουμε για αυτή τη νέα τάση που επικρατεί στην ε, Λατινική Αμερική και που επιχειρεί αυθαίρετα να αναθεωρήσει το σύνταγμα μια χώρα, διακόπτοντα την μέχρι τώρα παράδοση, παράδοση μίας ή το πολύ δύο θητιών προέδρων. Συνεχόμενων θητιών. Ήδη κάποιοι μίλησαν για άλλα τέσσερα θέματα. Σας ερωτώ λοιπόν, πότε πρόκειται να συζητήσουμε τα άλλα τέσσερα θέματα αφού μόνο τρία κατεπήγοντα επιτρέπονται. Ένα λεπτό δικαιούστε μόνο κύριε Κασουλίδη. Λυπούμε. Πρόεδρε, εγώ υποστηρίζω την άποψη της ομάδας μου ότι δηλαδή το θέμα αυτό δεν θα έπρεπε να είναι στην ημερησία διάταξη, γιατί υπάρχουν πολύ πιο επίγοντα και πιο σημαντικά θέματα διεθνώ. Εάν πρόκειται να εξετάσουμε την Ιχαράγωα, θα πρέπει να πούμε κιόλα ότι είναι μια χώρα που έχει τα υψηλότερα χρέη, μια από τις φτωχότερες χώρες Λατινικής Αμερικής. Αυτή την ε, τέος κομμουνιστική, το τέος κομμουνιστικό ε, πείραμα ούτε το φιλελεύθερο ε, πείραμα πέτυχαν. Είναι μια χώρα στην οποία ανακατεύτηκαν πάντα άλλες χώρες, η και άλλες. Και δεν έχει βγει καθόλου από την κατάσταση εμφυλίου πολέμου. Υπάρχει αυτή η τάση της σιδηράς Εμεί δεν θα πρέπει να το δεχτούμε αυτό, να το κατηγορήσουμε, αλλά υπάρχει παρόμοιο και στην ε, Ευρώπη. Κύριε Πρόεδρε, ελέγχθηκαν διάφορα. Καταρχήν ότι δεν είναι το σωστό θέμα γιατί υπάρχουν πιο επίγοντα θέματα όπου υπάρχουν περισσότερε καταπατήσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ίσως, αλλά εμεί ω Ευρωπαίοι που προσπαθούμε να τηρείτε το κράτο δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ελευθερία του τύπου, θα πρέπει να δούμε ότι κάπου απειλείται εδώ η ελευθερία αυτή και θα πρέπει να την προασπίσουμε. Ελέγχθη ότι το Ίδρυμα Φρίντριχ Νόμαν είχε συμμετάσχει στο πραξικόπημα Όχι, αυτό δεν είναι σωστό. Είναι φήμες αυτές και δεν μπορώ να το δεχτώ εξ ονόματος ε, του κόμματός μου. Μετά λέει το κύριο φαλάκη ε, αναφέρθηκε στο θέμα του προσωπικοποιήματος και γι' αυτό ε, απελάθη της χώρας. Μα άμα δεν πρέπει κανένας να συζητήσει ένα θέμα, τι γίνεται με την ελευθερία λόγου που έχουμε. Πώς μπορεί γι' αυτό να απελάσουν κάποιον απλώς επειδή συζητάει για οποιοδήποτε θέμα. Δεν έχει σημασία. Μα κοιτάξτε, δεν είναι αυτό ένα θέμα για απέλαση, νομίζω, μια λόγος για απέλαση επειδή συζητάει κάποιο θέμα. Αυτή δεν είναι καθόλου σωστή προσέγγιση. Ευχαριστώ κύριε Μάισνερ. Τελικώς, Τσάρλ Θάνοκ. Παραμένει η χώρα μια από τι πιο φτωχέ χώρε τη Αμερικανική Υπήρου και το ότι ο Ντανιέλ Τέγα δεν μπόρεσε να βελτιώσει την κατάσταση στη χώρα παρά από τόσε τόσε υποσχέσει σοσιαλιστικέ όταν ε, ανέλαβε την εξουσία σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνει αλλαγή φορά στην Νικαράγουα. Ε, το Σύνταγμα προβλέπει μία θητεία. Ε, πολλές φορές είναι η μακρότερη θητεία καλή για την σταθερότητα, όμως ε, εμπέζει το, το λαό, εμπέζει το κοινοβούλιο, έχει ευξημένες εξουσίες και κοιτάξτε τι έγινε και στη Βενεζουέλα με τον Ούγκο Τσάβες. Καουδίγιο όλοι κάνανε τον ηγέτη, τον ηγέτη της αριστεράς ε, όμως τελικά αυτή είναι η μεγαλύτερη απειλή για την σταθερότητα της δημοκρατίας και κοιτάξτε όλα τι γίνεται στη γειτονική τους ε, Ονδούρα, τι χάος βασιλεύει εάν πιστεύει σε ελευθερία και δημοκρατία τότε θα πρέπει κάτι να κάνουν προστατεύσουν τους πολιτέ της Νικαράγουας. Και ο κύριο είναι στο κατάλογο μου, παρακαλώ, ένα λεπτό. Ναι, πολύ σύντομα, πρόεδρε. Ένα αποτέλεσμα είχε αυτή η τόσο δύσκολη συζήτηση. Οι συνάδελφοι από τη Γερμανία της ομάδας ΑΛΔΕ επιβεβαίωσαν προηγουμένως ότι πράγματι το θέμα του πραξικοπήματος ήταν αντικείμενο των συζητήσεων αυτών. Το υπερασπίστηκε η συνάδελφος λέγοντας ότι μπορεί, πρέπει να μπορεί κανένας να συζητάει τα πάντα ακόμα και ένα πραξικόπημα. Μου φαίνεται ότι είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ε, αποτέλεσμα της συζήτησης και είμαι ευγνώμων γι' αυτό ευχαριστώ. Να τώρα την Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμοι συνάδελφοι, όπως γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ξεκινήσει αρκετά δύσκολο διάλογο με τη χώρα αυτή με στόχο την διαφύλαξη της δημοκρατίας και την ε, αποκατάσταση των δικαιωμάτων των πολιτών στα δημοκρατικά θεσμικά όργανα της χώρας. Επίσης, ε, έχουμε και τη μακροχρόνια δέσμευση να στηρίξουμε τη σταθερότητα και την ανάπτυξη όχι μόνο στη χώρα αυτή, αλλά στην ευρύτερη Κεντρική Αμερική. Μετά τις δημοτικές εκλογές του Νοεμβρίου του 2008, που στιγματίστηκαν από κατηγορίες εκταμένης νοθείας, η Διεθνής Διάσκεψη των Δωρητών ε, απέφθηνε κλίσεις που έμειναν ε, χωρίς συνέχεια. Η παραβίαση των δημοκρατικών αρχών και των ε, δημοκρατικών εκλογών ε, έφερε την ε, διάσκεψη των δωρητών να αναπροσανατολίσει τις δραστηριότητες συνεργασίας και να επανεξετάσει το πρόγραμμα ενίσχυσης προς τη χώρα αυτή. Η Επίτροπος Φερέρο Βαλτρίν αποφάσισε να αναστείλει οποιασδήποτε πληρωμές προς την Ικαράγου από την 1η η 2009 και μάλιστα τις της απόφασης προηγήθηκε συζήτηση με το Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη. Μετά από πολλαπλές επαφές με νοικουραγανές αρχές που έδωσαν δεσμεύσεις για πρόοδο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αρχές του Οκτωβρίου ε, κατέβαλε ένα εφάπαξ 10 εκατομμυρίων ευρώ από τον προϋπολογισμό υποστήριξης της Νικαράγουα για τον τομέα της παιδείας, κάτι που αποτελεί ένα απειροελάχιστο τμήμα των ε, κονδύλιο που έχουν ανασταλεί η καταβολή τους και που είναι 46 εκατομμύρια ευρώ. Μετά τις ε, εξελίξεις στο Συμβούλιο της περασμένης εβδομάδας ε, και επειδή δεν υπήρχαν προηγούμενες διαπραγματεύσεις με τα κράτη-μέλη, είναι πολύ σημαντικό όταν λαμβάνονται τέτοιου είδους αποφάσεις ε, να μην λαμβανονται αρων άρων-άρων αλλά να ακολουθείται μια διαδικασία που εξασφαλίζει ευθυγράμμιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά τη συμπεριφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι σε ένα κράτος, τρίτο κράτος. για να μπορέσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση να προβεί στα απαραίτητα διαβήματα. Η κυβέρνηση της Νικαράγωσης αποφα... ανήγγειλε ότι στις επόμενες δημοτικές εκλογές το 2010 και οι προεδρικές το 2011 θα μπορούν ε, να παρακολουθούν από διεθνείς παρατηρητές. Επίσης, ε, δεσμεύθηκαν να βελτιώσουν τον εκλογικό, τους εκλογικούς καταλόγους και να αποκαταστήσουν επαγγελματικές, εκλογικές και φορευτικές επιτροπές για το χρόνο. Βέβαια, Υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες για το κατά πόσο ε, είναι σοβαρές αυτές οι δεσμεύσεις και αξιόπιστες από την κυβέρνηση. Στις 21 Νοεμβρίου η Τρόικα εξέφρασε αμφιβολίες για τις τελευταίες εξέλιξεις στην Νικαράγουα. Η εφαρμογή όμως αυτών των δεσμεύσεων θα είναι, θα είναι αποφασιστική για την αναστολή της ενίσχυσης προς τη χώρα αυτή. Κάτι που θα αποφασιστεί μετά από διαπραγματεύσει και διαβουλεύσει με τα κράτη-μέλη. Γιατί δεν είναι μόνο θέμα που θα απασχολήσει μόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ολοκληρώνεται η συζήτηση για την Ικαράγουα. Η ψηφοφορία θα γίνει μετά το πέρας της συζήτησης και για τα τρία κατεπήγοντα. Συνεχίζουμε στο επόμενο θέμα. Έχουμε τέσσερα σχέδια ψηφίσματος για το Λάος και το Βιετνάμ και θα ήθελα να δώσω το λόγο στους